Και περνούμε αμέσως στην έκθεση του κυρίου Όλμπριχτ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση Πολωνία. Πρόκειται για μία μόνη ψήφο με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Le vote τη ψηφοφορία, όχι. Όχι λοιπόν, κρατούμε ακόμα ανοιχτή την ψηφοφορία για αυτή την πρώτη ε, ψηφοφορία. Le vote est clos. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Oui, on envoie un technicien pour votre machine, madame. Μάλιστα, σα στέλνουμε ένα τεχνικό για το μηχάνημά σα, ε, κυρία μου. Μισό λεπτό. Έκθεση Hoffman, ε, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Le vote. Avez-vous Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Et il est adopté. Εγκρίνεται. Le rapport de Monsieur Plenkovic. Plenkovic, έκθεση. Plenkovic, ονομαστική ψηφοφορία. Le vote. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Nous passons au rapport de Monsieur Negrescu. Έκθεση Νικολέσκου με ονομαστική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Έκθεση για την Μάκη. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Lightfried. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροποποιείται έτσι η θέση του Συμβουλίου. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Λαμασούρ. Τροπολογία 1. Ποια είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε για την πρόταση της Κομισιόν. Ποιοι είναι υπέρ, διανατάσεως της χειρός, ποιοι είστε υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Ζάλμπα Μπιντεγκάν. Τροπολογία 1. Δυνατάσιο της χειρός. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρόταση της, της Επιτροπής. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα το νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έκθεση Νηριάντα. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τώρα, για το ψήφισμα ε, με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Ταραμπέλα. Τροπολογία 1. Διανατάσεις χειρός υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 2 σε δύο τμήματα. τμήματα. Πρώτο τμήμα ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται. Μήπως μπορούμε να κάνουμε μια επαλήθευση παρακαλώ. Έλεγχος λοιπόν ηλεκτρονικός. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως έχουμε την ίδια πλειοψηφία, οπότε εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την παράγραφο 5. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία, εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την παράγραφο 9. Ψηφίζουμε. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για τη 10. Παράγραφος 10. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Διανατάσεις της χειρός για ε, την ε, τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 12. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, ίδια πλειοψηφία όπως πριν από λίγο, οπότε πιστεύω πως απορρίπτεται. Ελέγχουμε λοιπόν για το δεύτερο τμήμα της παραγραφού 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13, πρώτο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, παράγραφος 13. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές παρακαλώ επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 13 Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 14. Με ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 15 ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16 πάλι ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 20. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το επαληθεύουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 20. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Le Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Σε δύο τμήματα. Ποιο είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25, παράγραφος 25 σε δύο τμήματα, ε, πρώτο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, εποχές. Θα έλεγα πως εγκρίνεται, αλλά δεν είμαι βεβαία, οπότε κάνουμε παλήθευση. Για το δεύτερο τμήμα του 25 ψηφίζουμε παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 22. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ονομαστική ψηφοφορία για την παράγραφο 27 τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται περνάμε στην παράγραφο 28 ποιοι είναι υπέρ Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Παράγραφος 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 32. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 23. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται παράγραφος 39 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ονομαστική ψηφοφορία για την παράγραφο 41 άρχεται ψηφοφορία Τέλος της Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 και 17 που είναι ταυτόσιμες. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est clos. Et adopté. Εγκρίνεται. Nous passons au vote sur l'amendement 6 qui est Τροπολογία 6. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ξαναρχίζουμε γιατί δεν κατάλαβα. Ε, σηκώστε τα χέρια σα παρακαλώ. Υπέρ για την τροπολογία 6. Κατά αποχές να είναι πιο ξεκάθαρο τώρα εγκρίνεται 44 τώρα παράγραφος 44 ονομαστική ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται Περνάμε στην τροπολογία 11. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 46. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Je demande une minute. Ένα λεπτό παρακαλώ. Pardonnez-moi, il faut voter ναι, πρέπει να ψηφίσουμε για την τροπολογία 45. όντω. θα ψηφίσουμε λοιπόν για το πρώτο τμήμα της παραγράφου 45 με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Le vote clos. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, πάλι με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται Τέλος της πληροφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε στη 46, παράγραφο 46, ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην ψηφοφορία για τροπολογία 7. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την παράγραφο 49. Ε, ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την παράγραφο 50. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Ονομαστική ψηφοφορία για την παράγραφο 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 8 και 13 που είναι ταυτόσιμες. Σε ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζουμε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. στο τώρα τροπολογίες 9 και 14. Ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Le vote est Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Εκτιμώντας ε με διανατάσεις χειρός, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 19, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Εκτιμώντας η ε, ε, ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εκτιμώντας έλα ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στο εκτιμώντα σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στο εκτιμώντας R με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Έγκρινεται. Τροπολογία 20. Διανατάσσεως χειρός, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 15, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στο εκτιμώντας αε. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. Και περνάμε στο ψήφισμα, ε, στο σύνολό του, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Le vote ε, Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια, κύριε Ταραμπέλα. Και τώρα Nous allons passer euh, au vote. Nous allons passer au vote sur euh, le rapport de Monsieur Messerschmidt. Η έκθεση του κυρίου Messerschmidt τώρα, ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράγραφος δεύτερη, δύο τμήματα, διανατάσεως το πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται λέω τρίτο τμήμα ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει πέρασε εγκρίνεται δεύτερο ε, σε δύο τμήματα η τρίτη παράγραφος, πρώτο τμήμα υπέρ, δυνατά κατά. Απόχες εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, ονομαστικά υπέρ, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. απόχες, θα επαληθεύσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνώ τώρα στο δεύτερο τμήμα, διανατάσεως πάλι, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5, ονομαστική η ψηφοφορία, άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Ονομαστική ψηφοφορία για την παράγραφο 18 αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφο 40. Διανατάσεως υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη μάλλον. Ας επαληθεύσουμε όμως, αν το θέλετε. Παράγραφο 40. Επαληθεύουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 52 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 58 δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Παράγραφος 58. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 62 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές Εγκρίνεται μάλλον. 6. Τροπολογία 6. Αρχίζει ψηφοφορία ονομαστικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 διανατάσεως υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Ονομαστική ψηφοφορία για την παράγραφο 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 79 ονομαστική ψηφοφορία. Παράγραφος 79. Αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται παράγραφος 85, ονομαστική ψηφοφορία αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται παράγραφος 92 τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Παράγραφος 45 ονομαστικά αρχής ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7 ονομαστικά. Αρχίζει. Πέρας. Απερίφθη. Ε, παράγραφος 109 ονομαστικά αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. 117 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα ονομαστικά, αρχίζει. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά επίσης. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 2 ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Αιτιολογική σκέψη Β. Διανατάσσεως πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ψηφοφορία για την τρίτη παράγραφο ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 4 ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Το ψήφισμα ονομαστικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία για την τελευταία έκθεση της ε, συνεδρίασής μας. Έκθεση ζαλβα Μπιντεκαΐν. Τροπολογία 1. Διανατάσσος. υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Ονομαστικά παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και ευχαριστώ για τη συνεργασία